οι βουλευτές ε, Χουαν Κάρλος Βιντάλ και η κυρία Ινές Κριστίνα Τσούμπαρ ε, ανακοίνωσαν την παρέτησή του ως μέλη του Κοινοβουλίου από την 12η ε, Ιανουαρίου και 31η Ιανουαρίου αντιστοίχως. Το Κοινοβούλιο θα ενημερώσει τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Η Νομική Επιτροπή